και ελπίζω πως σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η τελευταία αιτιολόγηση ψήφου. Διακόπτουμε μέχρι τις 3.